και να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια για τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία Γιώρη. Περατώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Το επόμενο θέμα είναι η προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για ένα κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γκέρι, παρακαλώ τους συντάκτες της γνωμοδότησης, της ερώτησης μάλλον, ε, πρώτος ο κύριος Σταβαρές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρόσφυγες είναι ο πιο ευαίσθητος πληθυσμός, ο πιο τροτός πληθυσμός στον κόσμο, ιδίως όταν δεν μπορούν ούτε να γυρίσουν σε αιστείες τους, ούτε να πάνε σε άλλα μέρη. Η ανώτατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται σε 200.000 πρόσφυγες το χρόνο. Ε, η μισή από αυτού περίπου στον ΙΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Βραζιλία και Κίνα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρό ο πληθυσμό αυτό. Το Συμβούλιο έχει απαντήσει ήδη στο παρελθόν στην, στην ερώτηση αυτή. Η Σουηδία είπε ότι είναι έτοιμη να δεχτεί 5.000 περίπου το Βέλγιο λιγότερο, αλλά τονίστηκε από τις δύο προεδρίες ότι οι προσφύγες έχουν ένα ιστορικό δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τόνισε και η Ουγγρική Προεδρία ότι πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια εγκατάστασης των προσφύγων. Μετά από το 1956 ήδη τότε η διεθνή κοινότητα είχε ξεκινήσει την προσπάθεια επανεγκατάστασης των προσφύγων. Παραμένει όμως το δράμα των προσφύγων. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε αυτό το ερώτημα προς το Συμβούλιο. Πόσο μεγάλη προτεραιότητα για τα θέματα αυτά. Είναι τόσο μεγάλη προτεραιότητα ώστε τελικά να μπορέσει το Συμβούλιο να υπογράψει και να πραγματοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα αυτά η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, πηγαίνοντα από του Έλληνε κομμουνιστέ μέχρι του Βρετανού συντηρητικού, περιμένει από το Συμβούλιο να δράσει. Η διαδικασία λοιπόν τη ε, συναπόφαση δεν μπορεί να γίνει διαδικασία συν μη απόφαση. Θα ήταν ανόητο αυτό. Η έκθεση που εγκρίσαν εμεί αναφέρεται σε μέτρα κατεπήγοντα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση της ανθρωπιστικής αυτής κρίσης που αντιμετωπίζουμε και η οποία θα μπορούσε να συμβεί ανα πάσα στιγμή. Αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση προέρχεται από την Βόρεια Αφρική και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Δυστυχώ το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να περατώσει τη διαδικασία αυτή της συναπόφασης. Εμείς όμως πρέπει να βοηθήσουμε πέραν της ε, έκτακτης βοήθειας και τις χώρες οι οποίες θα πρέπει να βοηθήσουν στην επανεγκατάσταση των προσφύγων. Έχετε μόνο δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρος. Χρειαζόμαστε να υπάρχει μια πραγματική υποστήριξη προς τις χώρες αυτές οι οποίες επαναγκαθιστούν του ε, κλήρω, κύριε πρόεδρε, του πρόσφυγε. το Συμβούλιο, δεν πρόκειται εμεί να σα πούμε πώ θα λάβετε μέτρα, αλλά δεν μπορείτε εσεί να παραμείνετε σε αδράνεια. Συγγνώμη, πρέπει να σα διακόψω. Είχατε μόνο δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρο. Κλείνω, κύριε πρόεδρε. Χωρί μικρόφωνο μιλητή. Ο επόμενο ομιλητή, λέει ο πρόεδρο, είναι η κυρία Χίρς. Δύο λεπτά και εσεί έχετε πραγματικά δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Το πρόγραμμα επανακατάστασης ήταν ένα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ και εργαστήκαμε με πάρα πολύ πίεση και μας απορρόφησε πάρα πολύ ενέργεια σε όλες τις ομάδες. Στείλαμε ένα μήνυμα σαφές εφού συμφωνήσαμε και δώσαμε μεγάλη προτεραιότητα γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους. Ωστόσο παρά τις εξελίξεις ε, στη Βόρειο Αφρική, μάλλον λόγω των ε, περιστάσεων στη Βόρεια Αφρική θα πρέπει να εργαστούμε πολύ γρήγορα γιατί χάσαμε ένα χρόνο. Είχαμε το χρόνο και θα έπρεπε να τον έχουμε αξιοποιήσει για να κάνουμε κοινωνική συζήτηση στο ιστορικό της κοινωνίας γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξη των κρατών μελών, των δήμων, των κοινοτήτων, των περιφερειών Και αυτή η συζήτηση, αυτή η κοινωνική συνένεση η οποία αναπτύχθηκε κομμάτι-κομμάτι δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να δράσουμε σήμερα γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει και ως φιλελεύθεροι θα θέλουμε να θέσουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες συμφωνούν ότι αποστήλαμε ένα μήνυμα και τώρα αναμένουμε και από πλευράς του Συμβουλίου να δοθεί ανάλογη έμφαση, να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Τα άλλα κράτη-μέλη τα οποία ως τώρα δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό να συμμετάσχουν, να λάβουν κίνητρα. Ε, με από τον διάλογο ε, φαίνεται ότι υπάρχει προθυμία και από τα κράτη-μέλη. Άρα παρακαλούμε εμείς ως φιλελεύθεροι, αλλά νομίζω ότι συμφωνούν και οι υπόλοιπες ε, ομάδες, να θέσουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα να υπάρξει ευρεία κοινωνική συζήτηση και να μην υπονομευτεί αυτός ο διάλογος με την διαρκή αναβολή του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κυριος Παπανικολάου. Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζοντας τα όσα είπαν οι πολύ καλοί συνάδελφοι, να προσθέσω και εγώ τα εξής. Πρώτον, Κυρία Υπουργέ, ένα χρόνο σχεδόν μετά από τις αποφάσεις που εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο λάβαμε και πράγματι καταθέσαμε πολύ κόπο, πολλή προσπάθεια για αυτές τις αποφάσεις, κάναμε και αποστολή στη Συρία για αυτόν τον σκοπό και προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα προκειμένου όλο και περισσότερα κράτη μέλη να εμπλακούν στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων παρά λοιπόν όλα αυτά βρισκόμαστε ακόμη αδρανείς. και αν υπάρχει κάποιο τυπικό πρόβλημα από πλευρά συμβουλίου και πρέπει να εμπλακεί και το Κοινοβούλιο, εδώ είμαστε για να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Αναφερόμαστε στην ανθρωπιστική διάσταση του προγράμματος αυτού, αναφερόμαστε όμως και στο, στο μέσο που παρέχεται στην Ευρώπη για να ασκήσει ακόμη πιο αποτελεσματικά και εξωτερική πολιτική. Δεν θα ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό στα χέρια της κυρίας Άστον την περίοδο αυτή αν βρισκόταν στη Βόρειο Αφρική και μπορούσε να αναφερθεί και στο πρόγραμμα αυτό που θα είχαμε αποφασίσει. Βεβαίως αναφερόμαστε στις ανάγκες που υπάρχουν παγκοσμίω. Βεβαίως όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέον το πρόβλημα το έχουμε μπροστά μας. Η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη Μεσόγειο. Αυτό το πρόγραμμα κυρία Υπουργέ είναι απαραίτητο να το προχωρήσουμε, να το ξεκινήσουμε και πρέπει να αντιληφθούμε τη στιγμή που συζητάμε για τους δημοσιονομικούς πόρους μετά το 2013 ότι για το πρόγραμμα αυτό υπάρχουν αφιερωμένοι πόροι μέχρι το 2013 και αν χάσουμε και άλλο χρόνο δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους πόρους και αυτές τις δυνατότητες. Κλείνοντας κυρία Υπουργέ, θέλω να υπενθυμίσω την πρόταση που είχαμε κάνει και εκείνη την περίοδο και επαναφέρουμε διαρκώς σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό την, ομάδα μας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε σχέση με το πρόγραμμα εσωτερικής επανεγκατάστασης των προσφύγων, το λεγόμενο reallocation. Δεν μπορούμε, κυρία Υπουργέ, να περιμένουμε κι άλλες λαμπεντούζες να δούμε για να μπορέσουμε να δούμε την αναγκαιότητα και αυτής της πρωτοβουλίας που γρήγορα πρέπει να βάλουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. εντύμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο έχει τρία ερωτήματα από το Κοινοβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες των ερωτήσεων αυτών που ανέφεραν τις ιδέες που βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες αυτές ερωτήσεις. Τα τρία ερωτήματα αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός ταμείου για τους πρόσφυγες, την μεταρρύθμιση ε, του Ταμείου επίσης μεταξύ 2013-2015 στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος επανεγκατάστασης των προσφύγων. Το Κοινοβούλιο σίγουρα πιστεύει ότι η μοίρα των ανθρώπων αυτών των προσφύγων είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για την προσοχή που δείχνουν για την τύχη των προσφύγων και όπως είπε και ο κύριος Σταβάρης, έρχομαι από την Ουγγαρία, η οποία το 1956 γνώρισε ένα μεγάλο κύμα προσφύγων μετά την Επανάσταση του 1956 και αυτό μας δίνει και μια ιδιαίτερη ευθύνη να πάρουμε ένα ηγετικό ρόλο στα θέματα των προσφύγων. Η κρίση στη Βόρεια Αφρική, όπως είπατε, καταδεικνύει ότι χρειαζόμαστε μια ενιαία ρύθμιση, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των ρευμάτων προσφύγων. Και συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες τη για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, αν θέλουμε να παραμείνουμε σε ηγετικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων. το Συμβούλιο θα σας ε, δώσει και κάποια προπρόσφατα στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση στα σύνορα της Λιβύης. Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στα σύνορα της Λιβύης με την Τινησία όπου φτάνανε περίπου χίλιοι πρόσφυγες την ημέρα, ιδίω πρώην εργαζόμενοι στη Λιβύη που ζητούσαν να επαναπατριστούν, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν και υπήρχαν πολλοί από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν έγγραφα, δεν είχαν <clears throat> καθόλου ταυτότητες και έπρεπε να τους φροντίσουν οι διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές. Το πρόβλημα αυτό των ατόμων μπορεί να λυθεί μονάχα με μια διαδικασία ε, πανεγκατάστασης. Ο κύριος Μόρτουνη, Υπουργός Εξωτερικών, βρίσκεται τώρα στα ανατολικά σύνορα της Λιβύης <clears throat> με στόχο να αποκομίσει πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Ήρθε σε επαφή με προσώπους των Αιγυπτιακών αρχών και η κατάσταση έχει τροποποιηθεί. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται από τη Λιβύη προς τα Αιγυπτιακά σύνορα και προς το παρόν υπάρχουν 200 άτομα τα οποία είναι υποψήφια για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Τα υπόλοιπα άτομα τα οποία χρειαζόταν επανεγκατάσταση έχουν ε, εκενωθεί, έχουν ε, μετα... μετακινηθεί από τις Αιγυπτιακές Αρχές με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα και ο Σμορτούνη είναι σε επαφή με τον Υπουργό ε, εξωτερικών του Συμβουλίου της Φεγγάζης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου για να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Σε ό,τι αφορά την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τους πρόσφυγες, τονίζω ότι κάνουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και της δεσμεύσης μας για ένα κοινό σύστημα για τους πρόσφυγες το οποίο βασίζεται στο περιεχόμενο της Σύμβασης της Γενέβης του 1951 για το καθεστώς των ε, ε, προσφύγων και τις άλλες συναφείς διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Η Ουγγρική Προεδρία είναι δεσμευμένη για να προωθήσει τα θέματα αυτά που περιέχονται στο πακέτο για τους πρόσφυγες και επί τη βάση εντολής που μας έδωσαν τα κάτι μέλη είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον ε, άτυπο διάλογο για την οδηγία που αφορά τους πρόσφυγες με τα στοιχεία και να συλλέξουμε τα στοιχεία για το 2012. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που είχα την ευκαιρία να απαντήσω στα ερωτήματα του Κοινοβουλίου και θέλω να σας υπογραμμίσω ότι το Συμβουλίο αναγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος επανεγκατάστασης και έχει λάβει με ενδιαφέρον το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και την πρόταση της Κομισιόν από το Σεπτέμβριο του 2010 που ακολουθούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2008 για την παροχή ασύλου και την εθελοντική επανεγκατάσταση και αφορούν την επανεγκατάσταση στην Ευρώπη προσφύγων που βρισκόνται υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών. Η απόφαση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2008 επομένως έχει ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να επανεγκαταστήσουν πρόσφυγες στο εδαφός τους. Το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2009 ε, ενέκρινε και μία πρόταση για το Ταμείο των ε, προσφύγων, επανεγκατάσταση των προσφύγων και είχαμε και άτυπε συζητήσει το 2010 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη-μέλη έχουν δείξει μια ευέλικτη στάση έναντι των ε, προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρξει ένα πιο ευέλικτο καθεστώς για την επαγκατάσταση όπως τόνισε και η Κομισιόν. Όπως είπε και η Κομισιόν, ως αποτέλεσμα αυτών των ατύπων συζητήσεων μπόρεσε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πολιτικό, την πολιτική κατεύθυνση αυτών των προτάσεων. Και το Συμβούλιο υποστήριξε τη δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος θα ε, έδινε κίνητρα στα κράτη-μέλη με χρηματοδοτικά μέσα να προχωρήσουν στην επανεγκατάσταση των προσφύγων. Αλλά δεν μπορεί το Συμβούλιο να υποστηρίξει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το άρθρο 290 των συνθηκών και τις κατεχώρηση πράξεις για να δεχθεί μια διαδικασία πράξεων κατεχώρηση. Το Συμβούλιο εδώ συμφωνεί με την Κομισιόν θεωρεί ότι η διαχείριση του προγράμματος για τις μεταναστευτικές ροές θα πρέπει να γίνεται μέσα σε στενά χρονοδιαγράμματα και να υπάρξει αποτελεσματική σχεδίαση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Το Συμβούλιο φυσικά συμφωνεί και με την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι αιτήσιες προτεραιότητες για την επανεγκατάσταση αφορούν μονάχα εκτελεστικές εξουσίες. Δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μας επέτρεπε να έχουμε μια, ένα καθορισμό σε αιτήσιο επίπεδο των προγραμμάτων επανεγκατάστασης. Αλλά στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2013 έχουμε το ταμείο αυτό το οποίο υποστηρίζει την επανεγκατάσταση και ακόμα και σήμερα επί τη βάση των προτινομένων αλλαγών τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να έχουν ε, περισσότερη βοήθεια και να μπορεί να υπάρξει αναπροσδιορισμός των, ε, του αριθμού των προσφύγων και των περιοχών προέλευσή του. Αυτή τη στιγμή τα κρατημέλη μπορούν να πάρουν μέχρι 4.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα που επανεγκαθιστούν, ο οποίο εμπίπτει στι κατηγορίε οι οποίε έχουν συμφωνηθεί. Τίποτα δεν εμποδίζει τα κρατημέλη παρόλα αυτά στι τωρινέ συνθήκε να προβούν σε διαδικασίε επανεγκατάσταση που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα προγράμματα. Με χαρά σα αναφέρω ότι η Ουγγαρία από του χρόνου θα είναι τμήμα αυτού του προγράμματο και θα είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό επανεγκατάστασης. Και το Συμβούλιο παραμένει έτοιμο να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση η οποία θα έχει εφικτό χαρακτήρα και θα δίδει λειτουργικές και αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Η, η στόχη μας είναι, όπως αναφέρει και η πρόταση της Κομισιόν, η ευέλικτη χρήση αυτού του μηχανισμού και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού το θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν θα πρέπει να τύχει καθυστέρησης λόγω διαμαχών που έχουν νομικό χαρακτήρα. Τα θέματα των εκτελεστικών πράξεων έναντι των πράξεων κατεχώρηση, η σύνολη συζήτηση για τα θέματα αυτά έχει τροχοπεδίσει την έγκριση συμφωνίων για τα θέματα αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν πρέπει να καθυστερήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιώργη Και τώρα θα ε, έρθουμε στι πολιτικέ ομάδες. Ο κύριος Δίας Μέρα Γκαρφία. Το... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανείς δεν θα εκπλη... εκπλαγεί αν πω ότι η αλληλεγγύη με τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Δεν πρόκειται μονάχα για το θέμα αυτό, το θέμα της αλληλεγγύης με κοινωνίες οι οποίες είναι τροτές και ευάλωτες, αλλά έχει να κάνει και με τη γεωγραφική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται μια μεγάλη πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Η χώρα μου έχει αντιμετωπίσει πολύ έντονα τέτοια φαινόμενα, ενώ κάποιες άλλες χώρες έχουν υποστεί πολύ υποδέστερες πιέσεις. Καμία χώρα όμως δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα των προσφύγων. Επομένως, το πρόγραμμα για την ανα... επανεγκατάσταση των προσφύγων και τη χρηματοδότηση των κρατών μελών του 2010 δεν έχει περατωθεί ακόμα από το Συμβούλιο σε επίπεδο συναπόφαση. Τα λεγόμενα πολιτικά προγράμματα των κρατών μελών είναι μονάχα σταγόν εν το ωκεανό σε σχέση με το επίπεδο δράσεων που χρειαζόμαστε για την επαγγελματικατάσταση των προσφύγων. Οι χώρε του Νότου τη Ευρώπη αντιμετωπίζουν μια τεράστια πίεση, ιδίω μετά από τα λαϊκά κινήματα εξέγερση στην Αίγυπτο και την Τινησία και ο πόλεμο στη Λιβύα. Η <clears throat> Λαμπεδούσα με ένα πληθυσμό 5.000 κατοίκων έχει ε, υποδεχθεί ένα πολυπληθέστερο, πολύ πολυπληθέστερο πληθυσμό προσφύγων. Τα προγράμματα επανεγκατάσταση λοιπόν δεν μπορούν να ανακουφίσουν τη μεγάλη πίεση η οποία ισχύει σήμερα μόνο για την Ιταλία και τη Μάλτα, αλλά στο μέλλον θα έχει μια πολύ μεγαλύτερη έκταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τι χώρε αυτέ και είναι απαραίτητο το Συμβούλιο να ξεπεράσει τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη ενό προγράμματο επανεγκατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ξεπεράσει τι ε, μειοψηφίε εμπλοκή στο εσωτερικό του. Το θέμα αυτό τη επανεγκατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών αφορά το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μονάχα ένα τμήμα του την προηγούμενη εβδομάδα το ζήτησα και το ζητώ και τώρα να είναι παρόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα σύνορα της Λιβύης. Δεν είναι αρκετό το ότι πήγαν ορισμένοι συνάδελφοι στην Αίγυπτο. Πρέπει να είμαστε σε θέση από μόνοι μας να αξιολογήσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση και στη Λιβύη. Ευχαριστούμε κύριε Εκ Σοσιαλιστών Δημοκρατικών, λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Είναι σαφές ε, σήμερα ότι εδώ ε, διακομματικά υπάρχει το αίτημα από το Συμβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί να η επανεγκατάσταση των προσφύγων γίνει πραγματικότητα. Η επανεγκατάσταση των προσφύγων δεν σημαίνει μοίρασμα των βαρών. Πρέπει να βελτιωθεί το, σύστημα, το κοινό σύστημα αίτησης ασύλου. Αυτό που ζητάμε εδώ είναι να πέσουν τα εμπόδια που δημιουργούν δυσκολίες στο σύστημα επανεγκατάστασης στην Ευρώπη. Έχουμε 4.000 μόνο μετανάστες προβλέπετε. Αν δούμε τι γίνεται με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, συγκρίσιμα είναι τα μεγέθη. Μην ξεχνάμε ότι οι, οι περισσότεροι ε, που μετακινούνται στον κόσμο πάνε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε χώρες δηλαδή που δεν μπορούν να επομιστούν αυτό το βάρος η αξιοπιστία του συστήματός μας καλεί το Συμβούλιο να δράσει συνολικά για να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα επανεγκατάστασης. Αυτό συζητάμε εδώ μέσα σήμερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μωράης. Η κυρία Γκρίσμπεκ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ένα νούμερο πάνω από 10 εκατομμύρια πρόσφυγες στον κόσμο ευάλωτα άτομα, απειλούμενες γυναίκες, παιδιά, ανήλικοι, χωρίς συνοδό, σοβαρή κρίση. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση που να δείχνει ότι σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα. Μια διαπίστωση. Εδώ και ένα χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησε. Και ο συνάδελφος πιο πριν είπε το Συμβούλιο ας διαπιστώσει την ομοφωνία που υπάρχει στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και μια ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι είναι κοινικό το Συμβούλιο για να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή το ότι η πρώτη ανάγνωση δεν έχει προθεσμία και το έκανε αυτό για να μπλοκάρει τη διαδικασία συναπόφασης. Τι γίνεται με την επίγουσα επανεγκατάσταση, αυτή δεν μπορεί να περιμένει το 2012 κυρία Υπουργέ. Προτείνω να βγούμε από τη σχιζοφρενική κατάσταση που υποχρώνει τις χώρες μέλη να πάρουν σταθερές, στεναρές θέσεις στα λόγια, αλλά όταν Χρειάζεται το νομικό πλαίσιο, όπως εδώ, όταν υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη του σημερινού κόσμου, δεν γίνεται το ίδιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ένα λεπτό ο συνάδελφος Κίρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, μιλάω ως πρώην Υπουργό ε, Θεμάτων Μετανάστευση στη Μεγάλη Βρετανία. Δεδομένου των πρόσφατων γεγονότα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα που ε, υπόκεινται αυτού του είδου τι κινήσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε με εθνικά προγράμματα στο παρελθόν να καλύψει του μετανάστε. Πρέπει όμω με συντονισμένη προσπάθεια από κοινού να συζητήσουμε πώ είναι δυνατόν να συμφιλειώσουμε ένα σύστημα που βρίσκεται σε ανάγκε σε χώρε που έχουν τι δικέ του εθνικέ προτεραιότητε. Βέβαια, τα προγράμματα δεν θα υπονομεύουν τι εθνικέ αρχέ να παίρνουν αποφάσει. Επίση, χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Περισσότερο δράση και αποφασιστικότητα από το Συμβούλιο. Και θέλουμε να μα διαβεβαιώσετε ότι θα μα πληροφορείτε τακτικά περί του πρακτέου. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική επιταχύνουν τα πράγματα και αν αυξηθεί το βάρο, αν στο μέλλον αυτό σημαίνει στο υποχρεωτικέ ποσοστώσει ε, ε, μεταναστών ε, παρακαλώ πάρα πολύ το Συμβούλιο να δράσει άμεσα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Δυό Δυόμιση λεπτά η συνάδελφος Κουέλιο. Ευχαριστώ. Η επανακατάσταση είναι σημαντικό μέσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων. Όπως αναφέρθηκε, άλλες χώρες όπως η κάθε χρόνο επανακαταστούν ε, χιλιάδε. Ε, πρόσφυγες στην επικράτειά τους. Η επανεγκατάσταση είναι για τα άτομα τα οποία δεν έχουν προσπαθήσει να φτάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσουν άσυλο. Για άρα τα κρατημέλη λοιπόν που λένε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη μετανάστευση προτού έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέλειο εργαλείο. Ωστόσο υπάρχουν χώρες που είναι πολύ πιο φτωχές από τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλα αυτά ε, υποδέχονται πρόσφυγες όπως το Πακιστάν, η Συρία. Ωστόσο, επειδή αυτές οι χώρες δεν έχουν δυνατότητα υποδοχής, πολλοί πρόσφυγες ζουν σε απαράδεκτες ε, καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να βοηθήσει. Η επανεκατάσταση Ιρακινών προσφύγων κατέδειξε ότι λειτουργεί το σύστημα. Ωστόσο, ο αριθμός των Ιρακινών προσφύγων που έγινε αποδεκτός ήταν πολύ χαμηλός, γελία χαμηλός. Είναι απίστευτο το ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή προσπαθούν να εμποδίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του δικαιώματα και δεν είναι αποτεκτό να λέμε ότι η αναβολή, η καθυστέρηση της διαδικασίας αφήνεται σε εμά. Το Συμβούλιο καθυστερεί την διαδικασία γιατί δεν μας αναγνωρίζει τα καθήκοντά μας αλλά και τα δικαιώματά μας ως εκλεγμένοι του Ευρωπαϊκού Λαού. Άρα, ζητώ να μάθω το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που ε, έχουμε. Δεσμεύεστε προσωπικά να βάλετε το θέμα αυτό στην ατζέντα το συντομότερο δυνατό, γιατί χάνουμε χρόνο κάθε μέρα που περνάει. Και θα πρέπει να πω ότι εξετάζοντας και άλλα μέσα τα οποία έχουμε στην τρέχουσα κατάσταση και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Η επανεκατάσταση θα μπορούσε να μας βοηθήσει και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Βόρεια Αφρική. Μακροπρόθεσμα και άλλα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας που δεν χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, για την προσωρινή προστασία ή για την εσωτερική, ε, τον εσωτερικό διαμοιρασμό των προσφύγων. Δεν τα χρησιμοποιούμε και έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόθυμα δεν θέλουν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα, σας ρωτώ πώς σκοπεύετε να φροντίσετε ότι θα υπάρχουν κοινά συστήματα ασύλου μέχρι το 2012. Και Θεωρώ ότι είναι καθυστερημένο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Δεν ήρθε ο κύριος Μποργέζιο, άρα θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον συνάδελφο Σέγγιντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, μιλώντας για θέματα ε, μετανάστευσης σήμερα, προφανώς δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική και να τα αναλύσουμε. Κάτι που θα πρέπει να καλωσορίσουμε είναι ότι ο κόσμος αυτός πλέον σέβεται τη δημοκρατία, αλλά πολλοί κόσμος ε, χάνει τη ζωή του, άμαχος πληθυσμός, γυναικόπαιδα χάνουν τη ζωή τους. Και αυτό αποτελεί μόνο την βραχυπρόθεσμη απόρρια των όσων συμβαίνουν, αλλά θα υπάρξουν και μακροπρόθεσμες ε, συνέπειες. Σκεφτείτε τη Λιβύη, το μισό εκατομμύριο ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Και κάτι ακόμα που επιδεινώνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Η Δυτική Ευρώπη είναι έχει γεμίσει με πρόσφυγες. Η Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα άλλο πρόβλημα. Η μειονότητα των Ρωμά είναι ε, κυρίαρχη αναλογικά στον πληθυσμό και κοιτώντας τον αραβικό κόσμο ε, κυρίως πρόκειται για Αφρικανούς. Ας δούμε λοιπόν το εξής σενάριο. Αν αποδεχτούμε δεχτούμε την υποδοχή των ε, προσφύγων αυτών μπορεί να υπάρξουν εθνοτικές εντάσεις. Είναι αδύνατον με τη βία να επανακαταστήσουμε πιο πολλούς πρόσφυγες στην Ευρώπη. Να σας πω ότι η έννοια της μετανάστευσης είναι λανθασμένη. Κοιτάξτε, εδώ στην αίθουσα, πόσοι φιλελεύθεροι είναι εδώ στην αίθουσα συζητώντας ε, τα θέματα της μετανάστευσης. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ντρέπονται. Πώς πάλι να πετύχουν τους στόχους τους αν δεν είναι καν παρόντες σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι να δοθούν πόροι για τους ανθρώπους αυτούς εκεί που ζουν, στη Βορειοαφρική. Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή ήταν λοιπόν οι ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων και τώρα ο συνάδελφος Κοέλιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την κυρία Υπουργό να αναφέρει τη σημασία των προσφύγων και του προγράμματο επανεγκατάστασης. Τα στοιχεία του, της υπάτης αρμοστίας του ΟΗΕ είναι σαφή, μιλάνε για εκατομμύρια πρόσφυγες και 200.000 άτομα τα οποία κάθε χρόνο χρειάζονται επανεγκατάσταση. Υπάρχει μια ανθρωπιστική κατάσταση κρίσης στον σημερινό κόσμο. Δεν είναι μόνο το Αφγανιστάν, το Κονγκό, η Σομαλία, έχουμε την Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Λιβύη σήμερα αλλά πέραν από την ανθρωπιστική κατάσταση ε, ανάγκης, όπως είπε και ο κύριο παπα Παπα-Νικολάου, έχουμε και μια κατάσταση κονδυλίων του προπολογισμού που δεν μπορούν να δαπανηθούν γιατί δεν έχουν εγκριθεί τα προγράμματα αυτά. Άκουσα την κυρία Υπουργό επίσης να λέει ότι δεν μπορούμε για νομικούς λόγους να παραλύσουμε αυτή τη διαδικασία. Μα η διαδικασία έχει παραλύσει για λόγους ακριβώς νομικούς. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ε, συναπόφασης και βλέπουμε το Συμβούλιο να, να αντιτίθεται στις προτάσεις του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης το οποίο έχουμε διατυπώσει. Το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θέλει με νομικές ρυθμίσεις να εμποδίσει την έγκριση αυτής της αποφάσεως. Είναι ή δεν είναι σημαντικό για το Συμβούλιο το θέμα της επανακατάστασης των προσφύγων. Έχουμε το Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο και στη συνέχεια και ξέρει το Συμβούλιο ότι η πρότασή του σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα προέλευσης των, μεταναστών προσφύγων θα εξεταστεί μόνο το Ιούλιο. Δεν είναι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο καθυστερεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο ζητάει από το Συμβούλιο να αποφασίσει. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κουέλιο. Η κυρία Γκυγιόμ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, στα πλαίσια τη ανθρωπιστική κρίση στη Λιβύη, σήμερα περισσότερο από κάθε φλερά η Ευρώπη θα πρέπει να φροντίσει να δράσει συντονισμένα σε θέματα επανεγκατάσταση. Από την 1η Μαρτίου η διεθνή κοινότητα συμμετέχει σε μια προσπάθεια επανεγκατάσταση επιγόντω, αλλά Κανένα κράτο μέχρι σήμερα δεν δήλωσε την πρόθεσή του συμμετέχει στο πράγμα αυτό. Μόνο η Ιταλία πήρε μερικέ δεκάδε Ερυθρέου που φύγανε επιγόντω από την Τρίπολη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, μια υπόθεση επανακατάσταση 4.000 ατόμων μέσα στα πλαίσια του προγράμματο αυτού. Πείτε μα κάτι σχετικά. Η ευθύνη τη Ένωση ε, είναι σαφή και δεν πρέπει να επιτρέψουμε μη δράση. Χρειαζόμαστε αγγελεγγύη. Η Τινησία και η Αίγυπτος δέχτηκαν να ανοίξουν τα σύνορα σε αυτούς που φεύγουν από τη Λιβύη. Η Ευρώπη θα πρέπει να του υποστηρίξει και να λάβει το μερίδιό της στη διεθνή προστασία παροχής ε, βοηθείας στους ε, ε, μετανάστες, στους πρόσφυγες. Η Ένωση θα πρέπει πρώτη να έχει μια πιο γενναιόδρη πολιτική με την εγκατάσταση σε αυτούς για τους οποίους η τελική λύση είναι αυτό. Το 2009 400.000 πρόσφυγες επανεγκαταστάθησαν στον χρόνο αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό όμω από αυτού στα κράτη-μέλη τη Ένωση. Πέρα από τον προσωπικό αυτό στόχο, κάθε ευρωπαϊκή πολιτική επανεγκατάσταση θα πρέπει να φροντίσει για καλή προετοιμασία πριν φύγει ο υποψήφιο για την επανεγκατάσταση. Να καλύπτει κυρίω τα πιο ευάλωτα άτομα και να υπάρχει υποδομή υποδοχή. Τρίτον, συμπληρωματικά με τα εθνικά συστήματα ασύλου που υπάρχουν, η Ένωση θα πρέπει να έχει ένα σύστημα επανεγκατάσταση όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο που να στηρίζεται στις διάφορες εμπειρίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη με συγκεκριμένο συντονισμό. σε ευχαριστούμε κυρία Γκυγιόμ. Η κυρία Ρόσμπαχ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παντού σε όλο τον κόσμο έχουμε πολέμους, θεομηνίες και πρόσφυγες τα άτομα αυτά προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή. Περισσότεροι από αυτούς θέλουν να γυρίσουν στη χώρα τους. Πολλοί όμως είναι υποχρεωμένοι να επαναγκατασταθούν. Οι συνθήκε αλλάζουν συνεχώς. Λόγω των εντάσεων στη Βόρεια Αφρική η Ευρώπη έγινε χώρα σύνορο για χιλιάδες ε, πρόσφυγες και η πολιτική των κρατών μελών διαφέρει. Και ρωτώ, το Συμβούλιο μπορεί να μας πει αυτή η μεταναστευτική ροή τι θα σημαίνει σε σχέση με τα προγράμματα που εγκρίνονται στις Βρυξέλλες. Τα προγράμματα αυτά θα αυξήσουν τις κοινωνικές αρμοδιότητες σε θέματα ασύλου, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι και εγώ ερωτώ, το Συμβούλιο μπορεί να μας δώσει μια απάντηση, ένα χρονικό ορίζοντα διότι το Συμβούλιο θα πρέπει να μας πει είναι υπέρ ή κατά ενός ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης. Ευχαριστούμε. Σαφώς Ροπέρο Λόπες. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την κοινή γνώμη. Πώς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι είναι απαραίτητο να έχουν μια κοινή πολιτική επανεγκατάστασης. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να διατηρήσουν την κυριαρχικότητα για το θέμα του αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για να υπάρξει μια κοινοτική πολιτική, η οποία καθορίζει πολιτικέ και οι πολιτικέ θα πρέπει να αντανακλώνται στην κατανομή των κονδυλίων για του πρόσφυγε. Είναι απαραίτητο να υπάρξει λοιπόν μια λύση, γιατί υπάρχουν πολλέ δυνατέ λύσει. Το Συμβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την οδό. Αν τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση από το ταμείο αυτό χωρίς καμία προϋπόθεση δεν θα υπάρξει ποτέ μια κοινή πολιτική παραγκατάστασης προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή πολιτική ασύλου είναι μια πολιτική σε εκκρεμότητα. Δεν μπορούμε από αυτήν να εξαρτώμε την πολιτική για τους πρόσφυγες και δεν μπορεί η μοίρα χιλιάδων προσφύγων να εξαρτάται από αυτήν. Είναι απαραίτητο να δείξουμε συντονισμό και αλληλεγγύη για να μην υπάρχει περισσότερο βάρος για τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία φλασικό Φλασσικό-Βαμπένοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. αγαπητοί Προ... Ε, Υπουργέ, πριν από ένα χρόνο περίπου είπα εδώ στην αίθουσα αυτή ότι περίπου μισά μέλη της Ευρωπαϊκής ε, κράτη-μέλη έχουν ε, ε, προγράμματα επανεγκατάστασης. Δεν υπάρχει συντονισμός όμως μεταξύ των κρατινών μελών και γι' αυτό το κόστος της επανεγκατάστασης είναι πάρα πολύ υψηλό. Αν έχουμε πολιτική θέληση και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε προγράμματα επανεγκατάστασης βάσει αλληλεγγύης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο επανεγκατάστασης και το πακέτο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την, για την χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων όπου δεν υπάρχουν και για να υπάρχει κεντρική διαχείριση των δραστηριοτήτων. Είναι γνωστά τα περιστατικά και τα γεγονότα. Υπήρχε ε, πολιτική συνένεση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οριστικοποιήσει την πρόταση και να την καταστήσει προτεραιότητα. Ευχαριστώ κυρία Φλασίκο Βαμπένοβα και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων που έρχονται από πολέμους, ένοπλες συγκρούσεις, από καταστάσεις λοιμού, από την εκμετάλλευση των γυναικών και παιδιών που είναι θύματα λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων, χρειάζεται μια αλληλεγγύη για του ανθρώπου αυτού. Αυτό είναι ένα κεντρικό και ουσιώδε θέμα που απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα για τη βοήθεια των ε, προσφύγων για να βοηθήσει τις χώρες οι οποίες μαστίζονται ιδιαίτερα από τα προβλήματα αυτά που είναι κοντά στι χώρε προέλευση των προσφύγων η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική, οι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό απαιτούνται μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά και να ληφθούν κατεπηγόντω για να μπορέσουν να επανεγκατασταθούν οι πρόσφυγε με την αξιοπρέπεια που απαιτείται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αποφάσει οι οποίε καθυστερούν τη στιγμή που χιλιάδε άτομα χτυπούν κάθε μέρα την πόρτα μα και δεν παίρνουν καμία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φιγκερέντου. Η κυρία Γκάλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, όπως είπατε και υπογραμμίσατε, διαπιστώνουμε ότι τα πρόσφατα περιστατικά καταδεικνύουν ότι το θέμα των προσφύγων μπορεί να πάσα στιγμή να καταστεί θέμα έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερο κύμα μεταναστών στην Ευρώπη και δεν είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε στρατηγικά στην πρόκληση αυτή. Ένα από τα πιο βασικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι η επανεγκατάσταση. Φυσικά μπορούμε να ζητήσουμε καλύτερο συντονισμό και πιο πολύ αλληλεγγύη, αλλά χρειάζεται κοινωνική συνένεση σε πρώτη φάση. Και προς αυτήν την κατεύθυνση όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες. Χαιρόμαστε που η Ουγγρική Προεδρία δεν θέλει να άρει, δεν θέλει να ε, βάλει ε, νομικά εμπόδια για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Ευχαριστώ την ε, κυρία Γκάλ και τώρα ο, ο κύριος Όμπερμαϊρ κλείνοντας την διαδικασία Catch Ευχαριστώ Πρόεδρε μία μικρή ελιτιστική ομάδα θεωρεί ότι είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμός των προσφύγων στην Ευρώπη και ότι θα πρέπει να έρθουν και άλλοι πρόσφυγες επειδή είναι υψηλό το βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Αυτό είναι ιδιαίτερα περίεργο επειδή είναι χιλιάδες οι πρόσφυγες από τη Βορειοαφρική και είναι εκρηκτική η κατάσταση στην Λαπεντούζα στην Αίγυπτο και στην Τινησία θα πρέπει να αποφευθούν τα προβλήματα μάλλον ε, ε, ενσωμάτωση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και βιώσιμη βοήθεια που θα παρέχουμε προς τις δύο αυτές χώρες για να αποφύγουμε τα ρεύματα. Ευχαριστώ συνάδελφε Όμπερ Μάιερ και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκιόρη για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ε, πιο σοβαρές ερωτήσεις και θέματα. Καταρχήν, Α δούμε η Ένωση τι ιστορικό έχει. Πολλοί από εσάς είπατε ότι καθυστερούμε σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλε χώρε και ότι είναι πιο γενναιόδοροι από εμά. Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό. Αν δείτε τον αριθμό των προσφύγων φυσικά είναι λιγότερο από αυτούς που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Το Συμβούλιο προσπαθεί να βρει μια λύση μακρόπνοη για το πρόβλημα των προσφύγων. Δέστε πόσα αιτήσει υποβάλλονται στην Ένωση. Πόσε αιτήσει υποβάλλονται, επαναλαμβάνω. Είναι οι πιο πολλέ από ό,τι οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Και αναφέρω σε συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ του 27 στοιχεία, μεταξύ 2005 και 2009, όλε οι χώρε μα επαναλαμβάνω, είχαμε 1.150.000 τόσες χιλιάδες αιτήσει. Οι άλλες χώρες 300.000 τόσες αιτήσει για άσυλο. Δέστε τα δύο νούμερα. Τα νούμερα αυτά μιλάνε. Δεύτερο, πολλοί από εσά με ρωτήσετε για το χρονοδιάγραμμα της Προεδρίας μας. Είναι σαφές, πρέπει να σημειωθεί η πρόοδος, το θέμα επιγεί και το είπα αυτό και τον Ιανουάριο, όταν το πρόβλημα ήταν λιγότερο οξύ. γιατί, σε σχέση, δεν είχαμε τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική. Αλλά έχουμε συγκεκριμένα σχέδια και προσπαθούμε να επιταχύνουμε την κατάσταση. Η Βελγική Προεδρία προσπάθησε να προωθήσει στρατηγική για τον στόχο το 2012. Οι τέσσερι κανονισμοί για το Δουβλίνο, η οδηγία για την ε, εγκατάσταση μακράς διαρκείας, και άλλες δύο, και άλλες δύο οδηγίες, τέσσερις συνολικά, για την υποδοχή προσφύγων κλπ. Αυτή η στρατηγική υποστηρίχθηκε στο, και από τα τρία κοινοτικά όργανα και έδωσε αυτά αποτελέσματα. Τώρα η μακροπρόθεσμη παραμονή. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν και το Συμβούλιο θα εγκρίνει μετά από μερικές εβδομάδες επίσημα τη συμφωνία αυτή και την οδηγία για τα προσόντα. Η Ουγγρική Προεδρία έχει εντολή να ξεκινήσει ένα τριμερή διάλογο άτυπο. Θέλουμε να το αρχίσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται και υπολογίζουμε σε εσά ως εταίρο μας. Τέλος όσον αφορά τη Συμβουλία του Δουβλίνου. Σημειώθηκε πρόοδος στο Συμβούλιο, λίγα θέματα παραμένουν ακόμα εκκρεμή, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ πολιτικά για τις διαδικασίες και τους όρους για το υποδοχή προσφύγων. Η Κομισιόν έκανε δήλωση, είπε ότι θα κάνει νέα πρόταση. Πιο πριν η πρώτη ανάγνωση ε, της ε, ε, ε, οδηγίας αυτής ολοκληρώθηκε και στην Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών μελετώνται ενδεχόμενες τροποποίησεις της οδηγίας σε σχέση με τους πρόσφυγες. Οι δύο νομοθετικές αρχές μπορούμε να συμφωνήσουμε για το Eurodec ε, τη δήλωση για τη δήλωση του Δουβλίνου και με το που Κομισιόν θα μας κάνει την πρότασή της ή τις προτάσεις της μάλλον, θα συνεχίσουμε τη δουλειά. Βόρεια Αφρική. Ανάφερα όλες τις προσπάθειες της Ουγγρικής Προεδρίας. Την επίσκεψη στα σύνορα, στο Συμβούλιο στις 11 Απριλίου θα αξιολογήσουμε την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση αλλά για όσους από εσά μας επικρίνουν έχω να πω το εξής. Στα σχέδια πορισμάτων του Συμβουλίου αναφέρουμε το πόσο σημαντική είναι η κατάσταση των προσφύγων και αν το κρίνουμε αναγκαίο και ανάλογα με το ρυθμό προόδου θα συγκαλέσουμε και ένα έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στη διάρκεια του εξαμήνου μας Προσπαθούμε να επιταχύνουμε λοιπόν την νομοθετική δουλειά, κάνουμε ό,τι μπορούμε και θέλω και εσείς να κάνετε το ίδιο όπως επίσης και η Κομισιόν. Ο κύριος Κοέλιο και μερικοί άλλοι ανέφεραν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, την τροποποίηση του κανονισμού για τους πρόσφυγες. Είπα στην εισαγωγή μου ότι συμφωνούμε με το πολιτικό περιεχόμενο, είναι νομικό θέμα. Έχω μια νομική συζήτηση και μας έχει πιάσει κάπως όμοιρους. Αυτό συμβαίνει με όλα τα εργαλεία που έχουμε. Κάθε φορά συζητάμε για το αν θα είναι πράξεις που θα εφαρμόζονται άμεσα ή θα είναι χωρούμενες κλπ. Έχω λοιπόν να πω το εξή. Δέχομαι ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η νομική διαδικασία, η ακολουθητέα και είναι δύσκολο οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταλάβουν τι σημαίνουν οι η πράξεις εφαρμογής ή η εκχώρηση εξουσιών. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε λύση γρήγορα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Ταυτόχρονα πρέπει να τηρούμε και τη συμφωνία της Λισαβόνας. Αλλά η διαχωριστική γραμμή δεν είναι πάντα σαφής μεταξύ της των πράξεων εφαρμογής και των πράξεων που έχουν ε, που γίνεται ένα είδος πληρεξούσιος, μια εκχώρηση σε τρίτους. Ας το συζητήσουμε αυτό περισσότερο, ας διαπραγματευτούμε περισσότερο. Ένα πράγμα θέλω να ξανατονίσω. Ας μην πιανόμαστε όμοιροι από μια νομική συζήτηση. Στο Συμβούλιο του Ιουνίου θα βάλουμε θέματα των προσφύγων στην ημερήσια διάταξη. Ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της τρέχουσας κατάστασης. Αλλά πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο στην ημερήσια διάταξη και θα ακολουθήσουν πιο στεναρές αποφάσεις από ό,τι πριν από δύο ή τρεις μήνες. Υπήρξαν τώρα και άλλες ερωτήσεις, όπως τι θα συμβεί αν έχουμε ροές, μεγάλη ροή μάλλον προσφύγων. Πρέπει να κρατάμε τη φαντασία μας υπό έλεγχο. Υπάρχουν πολλές βαθμίδες στις διαδικασίες αυτές. Η Ένωση προσφέρει εξαιρετικό έργο έχουμε σχέση με τις αρχές της Ινησίας, την παγ, παγ, άλλες παγκόσμιες οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό, το πιο επίγον είναι ο επαναπατρισμός και αυτό συνεχίζεται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η επανεγκατάσταση δεν είναι επίκαιρο θέμα. Στην Ιταλία υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί. Η Ιταλία ήδη δέχτηκε 125 άτομα αν σημείωσα καλά το νούμερο τα κράτη-μέλη ενεργά λοιπόν παίρνουν μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε και ένα νέο νομοθέτημα. Το χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ και πάλι και για την προσοχή σας. Και όπως δήλωσε ήδη η Ουγγρική Προεδρία, θα αποδείξουμε ότι είναι μια Προεδρία με καρδιά και έχουμε και τη στρατηγική για τους Ρώμα. Ειδικά για τους πρόσφυγες θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους Ρώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν την πρόεδρο του Συμβουλίου. Ο κύριος Ταβάρης για διαδικαστικό θέμα. Όχι για να γίνει συζήτηση όμως. Μεθοδολογικό ερώτημα είναι αυτό. Μας είπε το Συμβουλίο ότι συμφωνούν με όλα εκτός από το άρθρο 290. Μετά από την συζήτηση με τους χειώδεις εισηγητές, θέλω να κάνω δύο μεθοδολογικά σχόλια. Κύριε Ταβάρες, έχουμε καθυστερήσει ήδη και δεν μπορώ να δεχτώ άλλα σχόλια πάνω στο θέμα της ουσίας Μόνο διαδικαστικές παρεμβάσεις μπορείτε να κάνετε. Πρέπει να